Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα όχι μόνο για λόγου ασφαλεία, αλλά και για να προστατεύσουμε του πιο ευάλωτου κρατούμενου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτό, στα πλαίσια όλων αυτών, υπέβαλα τι δικέ μου τροπολογίε για την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση και δίνω κάποια παραδείγματα για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι μηχανισμοί καταπολέμηση αυτή τη εξτρεμιστική και ακραία συμπεριφορά στα σοφρονιστικά ιδρύματα τη Ένωση. Συγκεκριμένα γίνεται σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει ε, την ε, μέθοδο ε, διαχωρισμού των κρατουμένων έτσι ώστε να αποφευχθεί η ριζοσπαστικοποίηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι εξτρεμιστές κρατούνται ξεχωριστά έτσι ώστε να αποφευχθεί η διάδοση εξτρεμιστικής προπαγάνδας ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους κρατούμενους των φυλακών για παράδειγμα απομάκρυνση εξτρεμιστικής, ε, ε, εξτρεμιστικού υλικού, κατάρτιση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης από το σοφρονιστικό προσωπικό κτλ. Θεωρώ πως αυτά τα μέτρα που έχουν ε, αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους τόσο στη χώρα μου όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέτρα τα οποία πρέπει να ε, διαδοθούν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και να πω επίσης ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας για να απομονώσουμε συγκεκριμένα περιστατικά σε κάποια χώρα. Τα σοφρονιστικά ιδρύματα έχουν πολλές ομοιότητες σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και δεν θεωρώ πώς θα ωφελήσει αυτή η πράξη απομονωτισμού ε, και παραδειγματισμού. Δεν νομίζω να καταφέρουμε ε, οτιδήποτε αποτελεσματικό με αυτή την ε, διαδικασία. Όμως ε, να πω πως χαίρομαι πως υπάρχει γενικότερη συνένεση ανάμεσα στους κοιόδης. Γι' αυτό λοιπόν στις επόμενες συνεδριάσεις είμαι σίγουρος πως θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά, όπως έχουμε ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν και θα οδηγηθούμε σε πολύ επικοδομητικές συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γέζεκ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι η γενικότερη προσέγγιση αυτής της έκθεσης είναι αρκετά ισορροπημένη. Η ομάδα μας ε, βάλε αρκετές τροπολογίες με στόχο να αντιμετωπίσει το θέμα του υπερπληθυσμού των φυλακών, της κατάρτισης ε, τόσο των κρατούμενων όσο και του σοφρονιστικού προσωπικού και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπή συνθήκες κράτησης ε, και διαβίωσης όχι μόνο για τους κρατούμενους αλλά και για το προσωπικό που εργάζεται στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Ο αριθμός των κρατούμενων έχει ξεπεράσει τις διαθέσιμες θέσεις σε ορισμένες φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο υπερπληθυσμός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στην προσπάθεια επίλυση αυτού του προβλήματο με επικοδομητικέ συστάσει, οι οποίε θα μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα, υπερπληθυσμός των ε, φυλακών έχει άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια και επηρεάζει αρνητικά τις ε, υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, το οποίο αποτελεί εμπόδιο γενικότερο για την κοινωνία. Σε γενικές γραμμές πρέπει να αρθούν τα εμπόδια και να υπάρχει επαρκής κατάρτιση των κρατούμενων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επανένταξή τους στην κοινωνία. Και με αυτόν τον τρόπο θα ε, αποφύγουμε και το θέμα του συνοστισμού. Επίσης, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα στις φυλακές. Γι' αυτό η κατάρτιση του ε, προσωπικού είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεται λοιπόν να στηρίξουμε την ε, κατάρτιση του προσωπικού των σοφρονιστικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα στην αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης. Πρέπει δηλαδή να, τους, ε, να δοθεί στο προσωπικό σοφρονιστικών ιδρυμάτων ε, επαρκής ε, εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να αποτρέπουν την ριζοσπαστικοποίηση. Χρειάζεται επίσης ίσως μια δημιουργία ενός κέντρου αριστείας όπου θα γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και θα υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε προσωπικό και σε κρατούμενους. Επίσης να τονίσω ότι πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των κρατούμενων ιδιαίτερα των ανήλικων, οι οποίοι θα πρέπει να κρατούνται ξεχωριστά από τους ενήλικες σε κάθε περίπτωση και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα. Υπάρχουν πάρα πολλέ φυλακέ στην Ευρώπη που ταιριάζουν πάρα πολύ στην περιγραφή του πρώην Υπουργού Ιστορικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος είπε ότι οι φυλακέ είναι ο καλύτερο τρόπο για να κάνεις τον κακό χειρότερο. Ελπίζω λοιπόν η εισηγήτρια και η σκιώδης να ε, συμπεριλάβει τις δικές μας απόψεις στην έκθεση και να την ευχαριστήσω καθώς και όλους τους σκιώδης για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρυσόγονος εκ μέρους της uh, this... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης στις φυλακές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ομάδα μας ε, GUNGL ε, τη βλέπει θετικά. Οι δικές μας τροπολογίες αποσκοπούν ε, στο να υπογραμμίσουν ειδικότερα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για παράδειγμα, διευκολύνοντας ε, τους ε, κρατουμένους να κρατώνται κοντά στα σπίτια τους ώστε να είναι δυνατή η επανένταξη στην κοινωνία και οι επισκέψεις από τους συγγενείς τους. Οι τροπολογίες μας επίσης ε, απαιτούν σωστή στελέχωση των φυλακών και καλές συνθήκες κράτησης, κάτι που είναι υποφελές για τους κρατουμένους. Η θέση μας όσον αφορά την έκθεση αυτή γενικότερα είναι θετική. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Ευχαριστούμε και για τους πράσινους. Τώρα η κυρία Ευαζολή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Συγήτρια, την κυρία Μπερζερόν για αυτή την έκθεση. Είναι αξιοσημείωτο ότι μία έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας συγκεντρώνει 284 τροπολογίες. Διαπιστώνω ότι είναι ευρία η συνένεση μεταξύ των ομάδων πέραν κάποιων εξτρεμιστικών ομάδων. Συμφωνούμε κατά τα άλλα όλοι στο να καταγγελούμε τις συνθήκες κράτησης, το συνοστισμό στις φυλακές, την ανάγκη οι φυλακές να γίνουν ένας χώρος επανένταξης και όχι απλά ένας χώρος ε, τιμώρησης. Την ανάγκη να υπάρχουν δραστηριότητες για τους κρατουμένους και να μην παραμένουν ε, άπραγοι για ολόκληρα 18 ώρα την ανάγκη ενασχόλησης με τα ευάλωτα άτομα και πρόσβαση σε υγειονομική περιθάλψη, η ανάγκη υλοποίηση εναλλακτικών ποινών, η ανάγκη διατήρησης των οικογενειακών δεσμών και η προστασία των συμφερόντων των παιδιών, η πρόληψη της υποτροπής, ε, η λήψη υπόψη των ε, συνθηκών εργασίας του συμφωνιστικού προσωπικού, εμείς ε, ως πράσινοι δεκρινόμαστε στο εξή. Θεωρούμε ότι πρέπει να εξετάσουμε αυτή την ιδέα της απομόνωσης των ριζοσπαστικοποιημένων. Σε πολλές χώρες επαναρχόμαστε σε αυτή την πρακτική. Είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης ε, αυτών των ατόμων. Πιστεύω επίσης ε, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε την αποποινικοποίηση της χρήσης της κάναβης ε, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των κρατουμένων. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και μια άλλη ιδέα που εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες ότι ένας, ε, σε κάθε νέο κρατούμενο θα αντιστοιχεί ένας νέος ε, αποφυλακισμένος. Και αυτή η ιδέα των ατομικών κελιών. πιστεύω ότι στην εκθέση αυτή θα καταφέρουμε να επιτύχουμε εύκολα συμβεβαστικέ ε, τροπολογίες και χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η η συγγήτρια δεν επιθυμεί να επανέλθει, θα ήθελα να την ευχαριστήσω αυτήν και τους Σκιώδης για την εντατική του συμμετοχή που είναι μεν ε, έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά όπως αποδεικνύεται ε, πολύ σημαντική λόγω του αριθμού των τροπολογιών. Θέλετε να μιλήσετε. Απλώς ήθελα να επισημάνω ότι όντω συμφωνούμε όλοι. Απλώς ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο θέμα ότι η ριζοσπαστικοποίηση μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, αλλά η ριζοσπαστικοποίηση επίσης συνδέεται με το συνοστισμό στις φυλακές και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ζουν στη φυλακή δεν έχουν άλλες, ε, όταν δεν έχουν άλλες ελπίδες, ε, η ριζοσπαστικοποίηση τους ανοίγει ένα παράθυρο επικίνδυνο μένα, αλλά ένα παράθυρο. Ο συνοστισμός λοιπόν και οι κακές συνθήκες διαβίωσης θα, θα έλεγα είναι η πηγή όλων των κακών. Και συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Ζολή, ότι το να απομονώνουμε τους ε, ριζοσπαστικοποιημένους ε, ε, δημιουργεί το κίνδυνο να τους ριζοσπαστικοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Καλύτερα είναι να εργαστούμε πάνω στους ανθρώπους αυτούς παρά να τους απομονώσουμε. Ε, είναι βασικό να υπάρχει κατάρτιση για τους ε, δεσμοφιλικές, για το σοφρονιστικό προσωπικό, γιατί αυτοί είναι αυτοί που θα εντοπίσουν τα πιο ευάλωτα άτομα που ε, είναι πιο πιθανόν να ριζοσπαστικοποιηθούν. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος και εσάς και όλους τους σκιώδεις. 21 ε, Ιουνίου θα γίνει η ψηφοφορία. Ε, περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην Ένωση. Στις 30 Ιουλίου ε, η Κομισιόν υπέβαλε το δεύτερο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει και ε, μία, στις 13 Ιουλίου συγγνώμη. η ε, πρόταση αφορά την αντικατάσταση της οδηγίας 2013 του κάθετος 32 και αφορά κοινέ διαδικασίες για την χορήγηση και απόσυρση της διεθνούς προστασίας στις 26 Ιουνίου του 2013 οι συντονιστές διορίσαν τη Λάουρα Φεράρα ως εισηγήτρια. Ε, έχει κάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις τους περασμένου μήνες με όλους τους ενδιαφερόμενους και είναι έτοιμη τώρα να μας ε, παρουσιάσει ε, το σχέδιο της έκθεσής σας και θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συναδέλφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε επικοδομητικά τους τελευταίους μήνες. Ήταν ε, σύνθετη δουλειά μας, πολύ τεχνικός ο κανονισμός και πολύ σημαντικός για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν στη διαθεσή μας διαρκώς. Κάναμε διάφορες συναντήσεις ε, για να εξετάσουμε άρθρο προς άρθρο ολόκληρο το κείμενο του ε, κειμένου του κανονισμού. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν για τη διαθεσιμότητά της και ευχαριστώ και όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, τους διαφορούς ενδιαφερομένους με τους οποίους ε, ήρθαμε σε επαφή όλους αυτούς τους μήνες και που μας προσέφεραν σημαντικές προτάσεις και ιδέες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους ε, με όσους ήρθαμε σε επαφή κατά την περίοδο που κάναμε σε διάφορα κρατή-μέλη στη Γαλλία, στη Σουηδία, στο Βέλγιο ήρθαμε σε επαφή με οργανισμούς, ε, οργανώσεις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές ε, σε διάφορα κράτη-μέλη προσπαθώντας να καταλάβουμε τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εκάστοτε χώρες να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να δούμε και ποιες ήταν οι απόψεις τους για αυτό το νομοθέτημα και ποιες ήταν οι συστάσεις τους. Αυτό που προέκυψε από όλες αυτές τις συναντήσεις είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται δίκαιη και ίση πρόσβαση στην, προστασία διεθνούς, στην διαδικασία διεθνούς προστασίας. Σωστή εξισορρόπηση μεταξύ του στήρισης των διαδικαστικών εχέγγυων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και από την άλλη της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Κάτι που συχνά δημιουργεί τάσεις και κοινωνικέ τάσεις στα κέντρα υποδοχής ε, ετούντων άσυλο ε, με αποτέλεσμα πολλές φορές ε, λόγω της αβεβαιότητας, της στασιμότητας των ετούντων άσυλο που συχνά πρέπει να περιμένουν ένα χρόνο πριν μάθουν ποιο είναι το νομικό τους καθεστώς, πριν μάθουν αν θα λάβουν ή όχι διεθνή προστασία. Από την άλλη αυτό συμπεριλαμβάνει και τεράστιες δυσκολίες για τα κράτη-μέλη που υποδέχονται τους ετούντε άσυλο δυσκολίες και οικονομικές, ε, διότι είναι δύσκολη η διασφάλιση επαρκούς και εξωπρεπούς υποδοχής για τα άτομα αυτά για πολλούς μήνες. Παναλαμβάνω λοιπόν, η σωστή εξισορρόπηση έγκυται στην τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των εχέγγυων αφενό, αλλά και τη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών με τη μείωση ταυτόχρονα του αναλογού κόστου. Πιστεύω λοιπόν ότι συμφέρει και τους του άσυλο και τα κράτη-μέλη οι αιτήσει να διεκπεραιώνονται εντό εύλογων χρονικών διαστημάτων. Κυρίως ε, οι αιτήσει που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν δεκτές, ε, που είναι σωστά θεμελιωμένες και τεκμηριωμένες ε, σε σχέση με τις άλλες που είναι αβάσιμες. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές που είναι βάσιμε θα πρέπει να διεκπεραιώνονται ταχύτερα. με σκοπό να μειωθούν και οι σχετικές δαπάνες. Είναι σημαντικό λοιπόν να διοχετεύουμε τις αιτήσει προς τη σωστή διαδικασία. Με τον κανονισμό αυτό λοιπόν έχουμε διάφορες διαδικασίες και είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε ποια είναι η σωστή ε, για τη διεκπαιρέωση των ε, επιμέρους ε, αιτήσεων ασύλου ανάλογα με τον τύπο τους. Θα πρέπει να γίνεται δηλαδή να εξετάζεται η κάθε αίτηση επί της ουσίας, να αξιολογείται κατά περίπτωση. Έτσι ώστε να προστατεύουμε διαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ έχω υποβάλει πολλές τροπολογίες. Τα βασικά σημεία της ε, έκθεσης ε, ε, αφορούν τη διαδικασία παραδεκτού, η εφαρμογή αυτή ήθελα εγώ να είναι ε, προαιρετική και όχι υποχρεωτική σε πολλά κράτη-μέλη μου υπογράμμισαν το ότι το να υπάρχει υποχρεωτική διαδικασία παραδεκτού αποτελεί ένα επιπλέον πρόσθετο βήμα το οποίο αντί να επιταχύνει τη διαδικασία την παρατείνει όλο και περισσότερο διότι απαιτείται ένα επιπλέον βήμα με το αναλογό κόστος φυσικά επιπλέον κόστος το οποίο θα πρέπει να υποστεί το εν λόγω κράτος μέλος. Οπότε σκόπιμο θα ήταν να παραμείνει προαιρετική. Μάλιστα η διαδικασία του παραδεκτού ε, δεν βοηθά την κατουσίαν εξέταση ε, του αιτήματο, οπότε και για την προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται πάντα επί της ουσίας εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Ε, με της, και πόσο μάλλον στις περιπτώσεις που, που αποτελούν εξαιρετικές περιπτώσεις Τώρα στις περιπτώσεις ε, ασφαλών χωρών καταγωγής θα μπορούσαν να γίνονται κάποιες ε, προληπτικές ε, διαδικασίες παραδεκτού. γιατί η διαδικασία παραδεκτού λοιπόν θα προτιμούσα εγώ να παραμένει προαιρετική και να μην υλοποιείται με τις έννοιες της πρώτης χώρας, ασφαλούς χώρας ασύλου ή, προ, ή ασφαλούς χώρας καταγωγής, γιατί δεν θέλουμε να αλλάξει το μοντέλο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Όσον αφορά την ε, ταχεία διαδικασία, από το κείμενο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται να είναι λίγο τιμωρητική η διαδικασία και η προσέγγιση αυτή. Εμείς, όπως είπα στην αρχή, θέλουμε να υπάρχει δίκαιη διαδικασία, να χρησιμοποιείται η σωστή διαδικασία για την ε, κάθε περίπτωση. Η ε, ταχεία διαδικασία λοιπόν μπορεί να χρησιμεύσει και στις περιπτώσεις όπου ε, υπάρχει ε, μια προφανώς ε, βάσιμη αίτηση. Αυτή η ταχεία διαδικασία λοιπόν μόνο, όχι μόνο σε περίπτωση αβάσιμης αίτησης αλλά και σε περίπτωση βάσιμης αίτησης. Έχουν αναφερθεί οι αναφορές της παραβιάσης των υποχρεώσεων του Δουβλίνου. Όλο αυτό γιατί, διότι είναι σημαντικό οι αρχές να έχουν ένα χρονικό όριο εντός του οποίου θα πρέπει να αποφασίζουν για τις αιτήσει αυτές αντί να αφήνουμε μια ακαθόριστη προτεραιότητα για τα αιτήματα αυτά. Εγώ έχω συμπεριλάβει δύο είδους ταχείες διαδικασίες, μία υποχρεωτική και μία προαιρετική. Η ε, υποχρεωτική θα μπορούσε ταχύες προέρχεται κάποιος από μια ασφαλή χώρα καταγωγής. Σε αυτή την περίπτωση ζητώ πλήρη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή ε, έναν ενιαίο κατάλογο χωρών ε, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Προαιρετική θα είναι η, διαδικασία, ε, η ταχεία διαδικασία στην περίπτωση αιτήσεων από τρίτες χώρες που θεωρούνται ασφαλείς ή από χώρες πρώτου ασύλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα την εφαρμόσουν ή όχι. Όσον αφορά τη συνοριακή διαδικασία, εγώ αποφάσισα ότι αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ποτέ στους ανηλίκους, είτε είναι συνοδευόμενοι είτε ασυνόδευτοι. Όσον αφορά τις διαδικαστικές συνέπειες λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων, εγώ ήθελα να μειώσουμε τις ποινές που προβλέπονται για τη μη τήρηση και την ε, αφαίρεση του ασύλου ήθελα τα κράτη-μέλη να μην, να μην τους επιβάλλεται κάποια υποχρέωση σε περίπτωση τέτοια. Τώρα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είπα στην αρχή, πρέπει να υπάρχει σωστή εξισορρόπηση μεταξύ της στήριξης των διαδικαστικών εχέγγυων και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρί να ξεχνάμε την αποτελεσματικότητα του συστήματο. Ειδικότερα θέλω να επισημάνω τρία σημεία. Πρώτον, να μειωθούν στο ελάχιστο οι περιπτώσει όπου μια ε, έφεση δεν δημιουργεί αυτόματα αναστολή. Διότι πέραν το ότι περιλαμβάνει τον κίνδυνο του ρεφουλμού και της ε, σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των ετούντων άσυλο, το να μην υπάρχει αυτόματη ε, αναβολή της έφεσης μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό για τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά θα δημιουργούνταν έτσι δύο παράλληλες διαδικασίες, μία που θα κινείται το επί της ουσίας για την έφεση και η άλλη για τη δυνατότητα του αν θα παραμείνει κανείς ή όχι στην επικράτεια αναμένοντας την εξέταση ε, της έφεσης, της προσφυγής. Αυτό λοιπόν θα οδηγούσε και σε κόστος που δεν μπορούν να αντέξουν τα κράτη-μέλη. Επίσης διαγράψα την δοκιμή της ουσίας ε, για το δωρεάν συνήγορο. Το γεγονό ότι έχει κανεί πρόσβαση σε ε, δικηγόρο από την αρχή της διαδικασία ε, βοηθά στην καλύτερη ποιότητα των αιτήσεων ε, με αποτελέσμα δεχομένω τη μείωση των περιπτώσεων έφεση. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται ότι από την αρχή θα υποβληθεί σωστά η αίτηση και συνεπώς βελτιώνεται η ποιότητα και της διαδικασίας καθώς και της προστασίας των θεμελιδών δικαιωμάτων. Ε, μετά για να είναι, πιο γρήγορες οι διαδικασίες έχω διαγράψει την μεταγραφή της ε, ε, ε, συνέντευξης, της ατομικής συνέντευξης. Αυτό το συζητήσαμε στη Γαλλία σε μια συνάντηση. Φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία ήδη εφαρμόζεται. Δεν μεταγράφεται δεν μεταγράφονται τα πρακτικά. Πραγματοποιείται μία οπτικοακουστική εγγραφή. Αυτό βοηθά στην προστασία των δικαιωμάτων για τους ετούντες άσυλο, οι οποίοι με αυτή την εγγραφή είναι σίγουρο ότι έχει καταγραφεί επακριβώς τα όσα, έχουν δηλώσει, αλλά βοηθά και στη μείωση του κόστους. Ε, πάμε να είναι απαραίτητο το, το άτομο που θα καταγράψει τα πρακτικά θα πρέπει να το μεταφράσει, θα πρέπει να γράψει μια περίληψη και ενδεχομένως να το ερμηνεύσει λάθος. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που σας παρουσιάζω τώρα περιληπτικά ε, και εύχομαι στη συνεργασία μας που θα συνεχιστεί με τους κοιοδησίτες να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό ε, ε περιληπτικό αποτέλεσμα. Ε, ένα ε, ικανοποιητικό συνολικό αποτέλεσμα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο που έχουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συζήτηση πρωτού περάσουμε στις τροπολογίες. Γι' αυτό θα ακούσουμε προσεκτικά τη γνώμη όλων των σκιωδών έτσι ώστε να αποκομίσουμε μια πρώτη εικόνα της κατάστασης. Ο σκιώδης του ΕΛΚ δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στο σκιώδη των Σοσιαλδημοκρατών, Πίτερ Νίντερμιλερ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την κυρία Φεράρα για, ένα, για μια εξαιρετική δουλειά, ένα πολύ δύσκολο θέμα. Όπως ε, αναφέρατε και εσείς, έχουμε εξαιρετική συνεργασία και θεωρώ ε, επίσης πως η Ευρώπη είναι έτοιμη να καταπιαστεί με αυτό το τόσο δύσκολο θέμα. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό που ήδη ανέφερε η κυρία Φεράρα, δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία στη διαδικασία και αυτή η διαδικασία να είναι ταχύτερη. Διότι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται είναι απαράδεκτη κατάσταση. Πολλοί πρόσφυγες περιμένουν 6, 8 μέχρι και 9 μήνες για την πρώτη τους ε, συνέντευξη. Δεν είναι δυνατόν. Είναι επίσης για μας πολύ σημαντικό αυτό που ήδη αναφέρθηκε, ότι δηλαδή κάθε αίτηση θα πρέπει να εξετάζεται ε, μεμονωμένα και ξεχωριστά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό θεωρώ πως χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, περισσότερη διερμηνία, περισσότερη πληροφόρηση στους πρόσφυγες και περισσότερα χρήματα ε, κατά επέκταση. Επίσης να πω πως ήδη γνωρίζουμε από τις συζητήσεις πόσο σημαντικός θα είναι ο ρόλος των προσφύγων στο μέλλον και συμμεριζόμαστε την άποψη της εισηγήτριας και επίσης θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να μην ε, προσπαθούμε να ε, δώσουμε έναν τιμωρητικό χαρακτήρα στη διαδικασία ασύλου, να μην τιμωρούμε τους ετούντες άσυλο αλλά να τους στηρίζουμε. Και να πω κάτι άλλο το οποίο ίσως ε, είναι κάπως αμφιλεγόμενο. Εγώ δεν συμφωνώ με τις αποφάσεις των κρατών μελών, διότι θεωρώ πως τα κράτη-μέλη προσπαθούν να επιλέξουν τον πιο εύκολο τρόπο, δηλαδή πώς να ε, διώξουν τους πρόσφυγες από το έδαφος τους. Χρειάζεται λοιπόν να συζητηθεί και ο ρόλος των κρατών μελών στην όλη διαδικασία. Ε, και να μην ξεχάσω να αναφερθώ στην ιδιαίτερη κατάσταση της Ιταλίας και της Ελλάδας. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάσουμε και αυτές τις διαφορές, αυτές τις ιδιαιτερότητες. Σε γενικές γραμμές πάντως στηρίζουμε την πρόταση στα κύρια σημεία της και θα ήθελα να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Φεράρα για το σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ. Ναι, η αντιπροσωπεία μας που πήγε στην Ιταλία και την Ελλάδα όντως ε, παρατήρησε χρόνους αναμονής μέχρι 9 μήνες. Και αυτοί οι χρόνοι αυξάνονται για την ομάδα ECR, ο κύριος Χαλά Άχο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα, ε, να ευχαριστήσω την κυρία Φεράρα για τη δουλειά τη. Νομίζω πω ε, δεν χρειάζεται να πω πως οι απόψεις μας διαφέρουν σε πολλά σημεία. Η ομάδα ECR είναι υπέρ της εναρμόνισης της νομοθεσίας για το άσυλο. Ο κύριος στόχος όμως αυτής της εναρμόνισης, κατά τη δική μας άποψη, θα πρέπει να είναι να αποθαρρύνουμε την παράτυπη μετανάστευση από τη μία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη τις ε, δευτερογενείς ε, ε, μετακινήσεις από χώρα σε χώρα. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι αυστήρη και όχι γενναιόδορη έτσι ώστε να εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Εάν υπάρχει αρκετή γενναιοδορία στα κοινά ε, πρότυπα, θα ενθαρρύνουμε την παράτυπη μετανάστευση. Βλέπετε τι γίνεται στη Μεσόγειο σήμερα. Πολλοί ε, που χρησιμοποιούν τη διαδικασία ασύλου δεν ε, χρήζουν πραγματικά προστασίας. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να έχουμε κοινά πρότυπα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι δευτερογενείς μετακινήσεις θα παραμείνουν πρόβλημα. Αυτό ισχύει για όλα τα σχετικά με το άσυλο θέματα τα οποία επεξεργαζόμαστε και έχουμε υποβάλει σχετικές τροπολογίες που ε, δείχνουν τη θέση μας. Γι' αυτό δεν χρειάζεται νομίζω να μπω σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεσίλη, εκ μέρους των Φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω, λέει κυρία Βίξτρομ, την εισηγήτρια για την εξαιρετική της έκθεση. Είναι ένα από τα δυσκολότερα θέματα στο χαρτοφυλάκιο του ασύλου. Σε γενικές γραμμές νομίζω πως είναι πολύ καλό να υπάρξει ένας κανονισμός που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της διαδικασίας αίτησης ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο προς ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ταυτόχρονα η εναρμονισμένη διαδικασία θα μας αναγκάσει να δώσουμε την ε, δέουσα προσοχή έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η αναγκαία ισορροπία που αναφέρουμε. Η διαδικασία ασύλου πρέπει να είναι γρήγορη αλλά ταυτόχρονα να ε, εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου. δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διασφάλιση ενός ε, εύρυθμου και λειτουργικού συστήματος δεν έχει να κάνει μόνο με το να τηρούνται οι προθεσμίες, αλλά και με την ασφάλεια δικαίου. Αυτό θα γίνει διασφαλίζοντας ότι οι αιτούντες άσυλο θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας και σε συνήγορο πολύ νωρίς τη διαδικασία αίτησης. Αυτό θα θα βοηθήσει έτσι ώστε η διαδικασία να μην είναι οικονομικά απαγορευτική. Και θα κατεβάσει το κόστος. Πρέπει να εξετάσω όλες τις προτάσεις της εισηγήτριας και να τις συζητήσω με την ομάδα μου. Θα ήθελα όμως ε, αρχικά να πω ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την εισηγήτρια. Η διαδικασία Αποδοχή μια αίτηση πρέπει να είναι προαιρετική για τα κράτη-μέλη. Και δεν θεωρώ πως υπάρχει λόγο στα κράτη-μέλη να αναγκαστούν να κάνουν κάτι αν ε, τα ίδια θεωρήσουν ότι η διαδικασία με αυτόν τον τρόπο θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Και κάτι άλλο. η απόσυρση της αίτηση ε, ασύλου είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Πρέπει να υπάρχει ρητή απόσυρση μιας αίτησης σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιος ε, δεν πηγαίνει στην προγραμματισμένη συνέντευξη, δεν τηρεί τις προθεσμίες που έχουν δοθεί. Αυτά βέβαια είναι λάθη ανθρώπινα. Γι' αυτό χρειάζεται κάποια ευελιξία. Εάν μια αίτηση αποσυρθεί ή θεωρηθεί πως έχει αποσυρθεί ρητά από τις αρχές, ο ετών δεν, θα έχει, δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επανυποβάλει αίτηση ασύλου και αυτή, σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια ε, επόμενη αίτηση που θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Βέβαια υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που, και ασφαλιστικές δικλείδες στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες όμως ε, είναι αρκετά δαπανηρές ε, και αφορούν την προσφυγή σε δικαστήριο. Υπάρχει μάλιστα μία διάταξη όπου μπορεί κάποιος να απελαθεί εάν οι αρχές θεωρήσουν μη παραδεκτή την ε, αίτηση ασύλου ή αν οι αρχές ε, θεωρήσουν ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία σε μία αίτηση ή αν κάποια αίτηση αποσυρθεί ακριβώς επειδή έχασε ένα ραντεβού για συνέντευξη ο ετών. σε περίπτωση που ασχηθεί έφεση από τον ετών, το πράγμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο και θα μας οδηγήσει σε μια καυκική ε, κατάσταση όπου ο ετών πρέπει να παραστεί αλλά δεν μπορεί να είναι παρόν γιατί τον έχουν απελάσει. Αυτό είναι πολύ περίεργο, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια θα μπορούσαμε να δεχτούμε να γίνεται μία έκθεση, μία αίτηση, να θεωρείται μία αίτηση πως έχει αποσυρθεί. Ρητά. Και αυτό σε περιπτώσεις όπου η άσκηση έφεσης θα είναι μια διαδικασία δαπανηρή και μακρόχρονη. Είμαι λοιπόν υπέρ της εναρμόνισης του συστήματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που χρειάζονται βελτίωση και εδώ είναι ο δικός μας ρόλος. Πρέπει εμείς να φροντίσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τη Λάουρα και το επιτελείο τους για την εξαιρετική τους δουλειά. Ευχαριστώ, Σίσιλη. Ε, υποθέτω ότι η συγγήτρια θα λάβει υπόψη σε αυτά που είπατε για τη σιωπηρή ανάκληση και κάποια άλλα θέματα που θίξατε. Η κυρία Άμπιο έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εργασία που ε, πραγματοποίησε η κυρία Φεράρα, η συγγετριά μας. Ε, είχαμε πολλές ευκαιρίες να ανταλλάξουμε ε, ιδέες και απόψεις με διάφορους οργανισμούς, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κυβερνητικούς φορείς και ήταν πολύτιμη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που είναι κατά της πρότασης της Κομισιόν γιατί απλώς παραβιάζει, θεωρούν, την Σύμβαση της Γενέβης υπάρχουν ε, διάφορες αντιρρήσεις ε, και αυτό ε, έχει ήδη γίνει κατανοητό αντιρρήσεις που αφορούν διάφορα σημεία της πρότασης της Κομισιόν. Και μέσω των τροπολογιών υπάρχει δυνατότητα να γίνουν βελτιώσεις και να απαλλαγούμε έτσι από όλα αυτά τα σημεία που αποτελούν παράβαση της Σύμβασης της Γενέβης. Τέτοια σημεία υπάρχουν σε διάφορες από τροπολογίες που έχουν έχουν υποβληθεί. Εμείς έχουμε κάποιες ερωτήσεις, ιδιαίτερα ε, σχετικά με το θέμα του μη παραδεκτού. των αιτήσεων ασύλου. Πότε θεωρούνται μη παραδεκτές οι αιτήσει ασύλου. Ε, θεωρούμε, ε, ιδιαίτερα αν ο λόγος είναι ότι ο ετών προέρχεται από μια ασφαλή χώρα, αυτό είναι ιδιαίτερα αμφίβολο, ε, γιατί είναι αμφίβολη αυτή η έννοια του τι είναι μια ασφαλή χώρα. Το να απορρίπτουμε δηλαδή αιτήσει ε, ασύλων από άτομα που προέρχονται από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση ή είναι ιδιαίτερα φτωχέ χώρες απλώς με βάση το επιχείρημα ότι είναι ασφαλείς οι χώρες αυτές, αυτή η ιδέα για μας είναι απαράδεκτη. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κατάλογος ε, των ασφαλών χωρών χωρίς να ξέρουμε με βάση ποια κριτήρια γίνεται αυτός ο κατάλογος, ποιος αποφασίζει ε, ποια χώρα είναι ασφαλής και ποια είναι όχι. Είναι ιδιαίτερα νεφελώδες το θέμα αυτό. Ε, για να βασιστούμε σε αυτό τι την έννοια ε, και να αποφασίσουμε για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας ε, ή καθεστώτος ασύλου. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν σαφείς ε, παράμετροι και σαφή κριτήρια για να καθορίζουμε, να αποφασίζουμε αν μια χώρα είναι ή δεν είναι ασφαλής. Ε, συμφωνούμε με διάφορες από τις προτάσεις που έχουν γίνει, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, νομική αρρωγή, ε, το χρονοδιάγραμμα, το ρόλο που παίζουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ιδιαίτερα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη της υπόλοιπη ομάδας, ε, ιδιαίτερα για το θέμα το, της λεγόμενης σιωπηρής ανάκλησης. Θεωρούμε ότι αυτή η έννοια δεν έχει καμία απολύτως νομική βάση. Είναι μια προσπάθεια ποινικοποίηση των ε, ε, ατόμων που υποβάλλουν αιτήσει και ελπίζουμε ότι θα απαλλαγούμε από την έννοια αυτή. Επίσης, η δυνατότητα απέλασης στη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής ή έφεσης, αυτή είναι μια ιδέα που είναι εντελώ ασύμβατη με οποιαδήποτε έννοια σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επίσης ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στον εντοπισμό των αδυναμιών ε, του συστήματος και επίσης ε, μιλάνε για μια σειρά εναλλακτικών ε, λύσεων για τη δημιουργία ενός συστήματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνάδει πλήρως με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ο σχεδόν ηγητής του ΕΛΚ έχει το λόγο. Ο κύριος Λενάρης, ευχαριστώ πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Είχαμε μια ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή. Και αυτή η διαδικασία θα πρέπει λίγα να απλοποιηθεί σε αυτό το κοινοβούλιο να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, όχι μόνο για την εκπόνηση της εκθέσης αυτής, αλλά και για όλες τις συναντήσεις ε, που διοργανώθηκαν. Ε, εξετάσαμε λεπτομερώς όλα τα άρθρα και ευχαριστώ και την Κομισιόν που διευκόλυνε την όλη διαδικασία. Αυτό βοήθησε όλους τους συναδέλφους και έδειξε επίση, ε, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, πόσο σύνθετη είναι αυτή η νομοθεσία και πόσο αναγκαίο είναι ό,τι κάνουμε εδώ να έχει συνοχή με όλες τις υπόλοιπες εκθέσεις και όλα τα νομοθετήματα που εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Το Κοινοβούλιο έχει πιστεύω τεράστια ευθύνη από αυτή την άποψη. Θα πρέπει να πάρουμε το ρόλο μας πολύ στα σοβαρά και να συνεχίσουμε την επικοδομητική μας συνεργασία. Θα είμαι σύντομος πιστεύω ότι ο κανονισμός ε, αυτός ε, βρίσκει σύμφωνη την Επιτροπή αυτή ως προς τους στόχους απλές διαδικασίες ε, με ίδια αποτελέσματα ανεξάρτητα από όπου υποβάλλεται μια αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω λοιπόν την πρόταση ορισμού των χρονοδιαγραμμάτων και των προθεσμιών για τα διάφορα βήματα της διαδικασίας αυτής, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσο εφικτά είναι αυτές οι προθεσμίες στην πρακτική. Διότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν ε, διαφορετικοί αριθμοί ε, μεταναστών ανάλογα με την περίοδο και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε το σύστημα που θα σχεδιαστεί εδώ να λειτουργεί καλά για όλα τα κράτη-μέλη σε εποχές χαμηλής και υψηλής ροής μεταναστών. Αυτό θα πρέπει να φαίνεται στι προθεσμίε που θα ορίσουμε. Επίση, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να μεριμνήσουμε για του ε, πρόσφυγε εκείνους που ε, προσπαθούν να ξεφύγουν από ε, τον πόλεμο και τη δίωξη. Αυτό σημαίνει ότι μια καλή διαδικασία επαναπατρισμού θα πρέπει να υπάρχει για όσου δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό ο κανονισμό να μην δώσει περισσότερα εργαλεία σε όσους ε, κάνουν αβάσιμες αιτήσει ε, χρησιμοποίηση της διαδικασίας και αόριστη παράταση τη παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, σε τελική ανάλυση μπορεί να χάσουμε και τα μέσα και τη δημόσια υποστήριξη. Και δεν θα μπορούμε πλέον να φροντίσουμε όσους πραγματικά χρειάζονται την προστασία μας. Θεωρώ ότι η έλεγχη παραδεκτού, η έννοια των ασφαλών χωρών και οι, οι διαδικασίες διαδικασίε διεκπαιρέωση θα είναι πολύ χρήσιμε έννοιε υπό αυτή την έννοια. Τέλο, να πω ότι όσον αφορά τα διαδικαστικά εχέγγυα και τι διαδικασίε για τα συνόδευτα ανήλικα, με πολλού συναδέλφου ε, πήγαμε στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα σε μια αποστολή τη Λίμπε. Συναντηθήκαμε με πολλά ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που έχουν κολλήσει αυτή τη στιγμή σε διαδικασίες σε διάφορα νησιά στην Ελλάδα. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά ένα 15χρονο κορίτσι από τη, που πήγε από την Αφρική στην Τουρκία με διακινητές ε, ε από τους οποίους ξέφυγε ε, στην Τουρκία γιατί την έβαζα να κάνει πράγματα που δεν ήθελε και τώρα έχει κολλήσει σε μια διαδικασία στη Λέσβο. Και είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται την ανάγκη μας. Τόσο πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πίσω στη Λόρα για τα συμπεράσματα. Συγγνώμη, η Κομισιόν θέλει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι από την ε, μονάδα ασύλου της ε, DG Home. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για, την, ε, για το σχέδιο έκθεσης της πρότασής μας. Προσμονούμε στην τελική έκθεση, η οποία πιστεύω θα αποτελέσει βάση για συζήτηση στη διάρκεια της νομοθετικής μας διαδικασίας. Να σημειώσω καταρχάς ότι συμφωνούμε με αυτό που τόνισε η συγκήτρια ότι δηλαδή πρέπει να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα της ε, διαδικασίας η οποία θα ωφελήσει τόσο τα κράτη-μέλη όσο και τους ετούντες άσυλο και τους εκπληκτές διεθνούς προστασίας, αλλά γι' αυτό θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό και το καλωσορίζουμε ότι αναφέρεται η επιθυμία να ε, συνεχίσει να χρησιμοποιείται η επισπρεσμένη διαδικασία. Και φαίνεται πως η εισηγήτρια συμφωνεί με την πρότασή μας ότι δηλαδή χρειάζεται να είναι σύντομο και λογικό χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης μιας ε, διαδικασίας αίτησης ε, ασύλου συμπεριλαμβανομένης και της έφεσης. Έχει δοθεί έμφαση στην έκθεση της εισηγήτριας, στην βελτίωση των δικονομικών δικαιωμάτων των ετούντων, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων, κάτι που θεωρούμε και εμείς αρκετά σημαντικό. Ιδιαίτερα μάλιστα δεδομένων των ε, μικρών χρονικών ε, περιθωρίων που έχουμε. Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση της όλης διαδικασίας ασύλου και να διασφαλίσουμε οι ετούντες ε, να κάνουν μία αίτηση η οποία θα εξετάζεται ξεχωριστά. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης κάποιες ανησυχίες, κάποια ερωτηματικά, ιδιαίτερα για το, για το πού θα εφαρμόζεται ο κανονισμός, αν θα μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα προξενείο μιας χώρας, ας πούμε. Νομίζω πως εδώ χρειάζεται αρκετή προσοχή για τις ε, για την πιθανότητα διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού εκτός της επικράτειας κάποιου κράτους μέλους. Επίσης, αναφέρθηκαν και κάποια άλλα σημεία από την εισηγήτρια, η δυνατότητα δηλαδή ύπαρξη κάποιων ε, διατάξεων που θα τροποποιούν την ερμηνεία του κανονισμού. Νομίζω πως ακούσαμε και από τους ε, σκιώδεις εισηγητές και από την εισηγήτρια ότι είναι πολύ σημαντικό να εναρμονιστεί η νομοθεσία στην Ένωση. Και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις ε, διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και να οδηγηθούμε σε μια πραγματικά κοινή διαδικασία ασύλου. Αυτές οι διατάξεις ενδεχομένως υπονομεύσουν το στόχο μας. Μετά, ε, η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και της χώρας αίτησης ασύλου είναι πολύ σημαντικές για την Κομισιόν. Η συγγήτρια έχει προτείνει να υπάρχει ένας προαιρετικός ε, χαρακτήρας ε, σε παραδεκτές αιτήσει αντί για υποχρεωτικό. δεν συμφωνούμε με αυτήν την πρόταση, ακριβώς γιατί το σκεπτικό πίσω από την ε, ασφαλή τρίτη χώρα είναι, έχει να κάνει με το αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφορά κάποιον που κάνει αίτηση ασύλου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν είναι απόλυτα σαφές για εμάς το πώς μια επισπεσμένη διαδικασία ε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί εδώ. Γιατί όταν ένα κράτος μέλος εξετάζει μια αίτηση, η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας δεν μπορεί να έχει κάποια εφαρμογή εδώ. Γι' αυτό θεωρούμε πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Και να σημειώσω κάτι άλλο η συγγήτρια προτείνει την ανάκληση κάποιων, κάποιων ε, λόγων επιτάχυνσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ε, επόμενων αιτήσεων. Τόσο στο διοικητικό αρχικό στάδιο, όσο και στο στάδιο της έφεσης. είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, υπάρχει μεγάλη σαφήνεια, ιδιαίτερα και στην περίπτωση των επιστροφών. Και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται επιστροφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως είναι σημαντική αυτή η επισπεσμένη διαδικασία ακριβώς για την ε, δρομολόγηση των επιστροφών ατόμων που έχει αποδειχθεί ότι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας και έχουν κάνει επανειλημμένα αιτήσει. Επίσης, η ανάκληση μιας έφεσης είναι και αυτό ένα ε, κάπως προβληματικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι ε, ο μη ανασταλτικός χαρακτήρας μιας αίτησης δεν ε, μπορεί να αλλάξει μια απόφαση. Δηλαδή, όταν κάποιο κάνει αίτηση και αυτή απορριφθεί σε διοικητικό στάδιο, θα πρέπει μετά να προσφύγει σε δικαστήριο, έτσι ώστε το δικαστήριο να αποφανθεί για το αν έχει δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα. Και το δικαστήριο λοιπόν εξοφίσει ο αποφασίζει Σε περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει επαναπροώθηση, τότε ε, θα χορηγείται το δικαίωμα της ε, παραμονής, της προσωρινής παραμονής. Τέλος, να πω και κάτι για τις επακόλουθες αιτήσει. Το καθεστώς της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συμφωνεί και με το κοινοτικό κατεστημένο μέχρι τώρα, θεωρεί πως η ανάκληση αυτής της ε, επιτάχυνσης βάζει σε κίνδυνο την όλη διαδικασία και την διαδικασία εξέτασης της αίτηση ασύλου σε διοικητικό στάδιο αλλά και στο στάδιο της Έφεση. Όταν έχουν γίνει πολλέ επακόλουθες αιτήσει μόνο και μόνο για να καθυστερήσουν την επιστροφή του ατόμου, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ε, ταχείας έτσι ώστε οι υπηρεσίε ασύλου να μπορούν να ασχοληθούν με άλλε αιτήσει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Προεδρία του Συμβουλίου, η Προεδρία της Μάλτας, παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Φεράρα και τους Σκιώδης για την δουλειά τους και γενικά την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όπως όλοι ήδη έχουν τονίσει, το θέμα αυτό χρειάστηκε ε, να γίνει, απέτησε να γίνουν πολλές διαβουλεύσεις ε, μεταξύ των κρατών μελών. Ε, το σχέδιο αυτού του κανονισμού είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση λόγω της πολυπλοκότητας της πρότασης. Κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας συζητήθηκαν ε, συμβαστικές προτάσεις για τα άρθρα αυτά που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο σε μια πιο θεματική προσέγγιση, κυρίως ε, περιορισμός των καταχρήσεων και των δευτερογενών ε, κινήσεων, ε, διατάξεις που σχετίζονται με τους ετούντες με ειδικέ ανάγκες, ε, ασυνόδευτη ανήλικοι, ιατρικές εξετάσεις ε, και το ίδιο και για τους ε, ε, συνόδευτους ανηλίκους. Ήταν πολύ δύσκολα όλα αυτά τα θέματα όσον αφορά την κατάληξη σε μια συνεκτική πρόταση. Οι τεχνικές συζητήσεις για τα άρθρα αυτά συνεχίζονται στην ομάδα εργασίας για το άσυλο αυτή τη στιγμή. Φυσικά η Προεδρία μας πλησιάζει στο τέλος της, τέλος Ιουνίου και θα λάβει τη συνέχεια η Προεδρία της Εστονίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα γυρίσω τώρα στην ε, ε, Λάουρα Φεράρα για τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα ε, όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και για τις σημερινές τους παρεμβάσεις αλλά και για τη συνεργασία μας μέχρι τώρα. Επαναλαμβάνω ότι η πιο σημαντική πρόκληση θα είναι να διασφαλίσουμε την εξισορρόπηση και το σεβασμό των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων από μια μεριά και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αφετέρου. Κάτι που δεν είναι εύκολο γιατί πολλές φορές ε, η εξισορρόπηση αυτή μπορεί να λείπει ε, και να επιταχύνονται οι διαδικασίες εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των εγγυήσεων της διαδικασίας. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Ε, θέτοντας λοιπόν ως στόχο καταρχάς την εξασφάλιση αυτής της εξισορρόπησης, ε, με αυτό έχοντας ε, κατά νου έκανα τις τροπολογίες που σας παρουσίασα. Απαντώντας στις ερωτήσεις που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιες μικρές παρατηρήσεις. Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας και η έννοια της πρώτης χώρας, ασφαλούς χώρας ασύλου, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαδικασία παραδεκτού, γιατί η διαδικασία παραδεκτού αποκλείει την εξέταση επί της ουσίας. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να αξιολογήσουμε ανά περίπτωση, αν πραγματικά η τάδε τρίτη χώρα ή η τάδε χώρα διέλευσης ε, πραγματικά ε, διασφαλίζουν για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, Πρόκειται λοιπόν για μια ε, αναπερίπτωση εξέταση που δεν ε, αποκλεί την διαδικασία επί ουσίας. Μπορεί να, να αποφασίσουμε για μια ταχεία διαδικασία, δηλαδή ένα κράτος μέλος να έχει μια λίστα με τις ασφαλείς τρίτες χώρες. Αλλά από εκεί και πέρα το να ε, οδηγηθούμε στην διαδικασία του παραδεχτού πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα υπονομευθεί αυτή η εξισορρόπηση, αυτή η ισορροπία που ε, στην αρχή και ότι θα επιταχύνουμε τη διαδικασία εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όσον αφορά το γεγονός ότι ανάμεσα στις τρεις περιπτώσεις ε, για την ταχεία διαδικασία αφαίρεσα την υποβολή της αίτησης μόνο με το σκοπό της ε, καθυστέρησης της επιστροφής αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πλατιά ερμηνεία. Ε, είναι πολύ ασαφής ε, ε, η διατύπωση αυτή, η έννοια αυτή και μπορεί να δώσει λαβή σε πολλές και διάφορες ερμηνείες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ένας κανονισμός πρέπει με μεγάλη σαφήνεια, εφόσον είναι ένα κανονιστικό κείμενο, να λέει ποιες είναι οι περιπτώσεις που με βεβαιότητα οδηγούν οδηγούν σε μια συγκεκριμένη διαδικασία και ποιε όχι. Η διακριτική ευχέρεια ε, που μας ε, ε, δίνει ε, αυτό το επιχείρημα ότι η αίτηση υποβάλλεται μόνο με σκοπό την καθυστέρηση δεν μπορεί να περιλαμβάνεται σε ένα κανονιστικό κείμενο. Ο, ο αυτόματος ανασταλτικός χαρακτήρας, το είπα στην παρουσίασή μου, το επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μας, το να περιμένουμε να υπάρξει μια διαδικαστική απόφαση που να αποφασίζει κατά πόσον, κατά τη διάρκεια εξέτασης έφεσής του, ο ετών άσυλο πρέπει να μείνει στη χώρα αυτή ή να γυρίσει στη χώρα καταγωγής του, αυτού μας φαίνεται ότι είναι μια τρέλα. Και από οικονομική άποψη, ε, όσον αφορά το οικονομικό βάρος για το κάθε κράτος μέλος, γιατί αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει ε, να επιστραφεί στη χώρα καταγωγής του το άτομο αυτό ε, και να υπάρχει περίπτωση να πρέπει να το ξαναφέρουμε στη χώρα υποδοχής εφόσον ο ετών άσυλο ε, αποφασιστεί ότι μπορεί να παραμείνει στο ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της προσφυγής του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβλέψουμε επίσης μια επιπλέον διαδικασία παράλληλα με την εξέταση της προσφυγής που θα αφορά τον ανασταλτικό χαρακτήρα. Από άποψη λογικής, από άποψη οικονομική, από άποψη θεμελιωδών δικαιωμάτων μας φαίνεται ότι είναι κάτι το παράλογο. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο υποβάλαμε αυτή την τροπολογία. Όσον αφορά τέλος, την δυνατότητα να εφαρμόσουμε ε, τον κανονισμό στα προξενία των κρατών μελών. Τα προξενία των κρατών μελών είναι έδαφος των κρατών μελών. Γι' αυτό δεν βλέπουμε για ποιο λόγο να μην μπορεί να ε, εφαρμοστεί και εκεί αυτός ο κανονισμός. Αντίθετα, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρω... επικράτεια των κρατών μελών ε, και ε, της Ευρωπαϊκής ένωση των κρατών μελών, άρα και στα προξενία των κρατών μελών, ε, που είναι, σύμφωνα με όλους τους κανόνες, έδαφος των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε πολύ, Λόρα απίστευτα σύνθετο θέμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είχαμε τη συζήτηση αυτή με τους Χιώδης και ότι υπάρχει καλή συνεργασία, όπως είπε και ο κύριος Λέναρτ, έχει γίνει πολλή δουλειά και με την Κομισιόν. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο η εναρμόνιση. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη συζήτηση. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 13 Ιουνίου. Για αυτό το λόγο το θέσαμε αυτό το θέμα ως θέμα προτεραιότητας. Είναι τα δυσκολότερα που έχουμε. Ευχαριστούμε για το, τις σας και εσάς και τους ε, σκιώδεις ε, και αναμένουμε τις τροπολογίες. Ας περάσουμε στο σημείο 11. Είναι το θέμα για την μετεγκατάσταση. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Η Μάλιν Μπιόρκ η συγκήτρια εισαγωγικά να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η πρόταση ε, εξετάζει την ανάγκη ασφαλών και νόμιμων αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει των ε, υπαρχουσών πρωτοβουλειών επανεγκατάσταση και ανθρωπιστική υποδοχή στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, καθώ και στην εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέσω των εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάσταση, ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ενωσιακό επανεγκατάσταση για να διευκολυνθεί η ενωσιακή πολιτική. 431 τροπολογίε έχουν υποβληθεί από τα μέλη να ζητήσω από την κυρία Μπιόρκ, την εισηγήτρια, να μας παρουσιάσει τις απόψεις της για τις τροπολογίες. Μάλλον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδους μου που βρίσκονται εδώ σήμερα και όσους δεν βρίσκονται εδώ, οι κατηπήροι ο Λιμισελ και η Χέλγα Στίβενς. Οι περισσότερε τροπολογίε φυσικά προέρχονται από του Κιώδη, αλλά και άλλοι συμμετείχαν. Θέλω να του ευχαριστήσω όλου γι' αυτό. Πριν από ένα μήνα, όταν παρουσίασα το σχέδιο έκθεσή μου στην Επιτροπή αυτή, ένα από τα βασικά μου σημεία ήταν ότι η επανακατάσταση εξχεδιασμού προστατεύει και παρέχει μια ασφαλή δίωδο και μια βιώσιμη λύση για τους ε, πρόσφυγες. Βασικός μου στόχος ε, ήταν δύο πράγματα να ε, διατηρηθεί η ανθρωπιστική ε, φύση της επανεκατάστασης και να αυξηθεί η επανεκατάσταση στην Ένωση. Και με χαρά μου βλέπω ότι οι τροπολογίες που έχω λάβει κινούνται ε, στην πλειοψηφία τους προς την ίδια κατεύθυνση. Η δημιουργία ενός φιλόδοξου πλαισίου επανεγκατάστασης βάσει ανθρωπιστικών αναγκών με αύξηση των αριθμών και συμπλήρωση της ε, υπάρχουσας ε, δομής επανεγκατάστασης διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει σημαντικότερο ρόλο στην επανεγκατάσταση παρέχοντας ε, ασφαλές οδούς για τους πρόσφυγες. Μέσω του τροπολογιών θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα για το περιεχόμενο που επιθυμούμε. Όσον αφορά τις τροπολογίες, ο βασικός ρόλος της UNHCR παραλαμβάνεται από πολλού Η ανθρωπιστική ουσία και φύση της επανεγκατάστασης, όπως είπα, ενισχύεται με τις ε, τροπολογίες και δεσφαλίστε μέσα στα άρθρα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Είχαμε φιλόδοξες τροπολογίες για την αύξηση των αριθμών και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το ε, δίκαιο μερίδιο διεθνούς ευθύνης. Σε διαδικαστικό επίπεδο είναι σαφές ότι διάφορες κοιόδες έχουν καταβάλει προσπάθειε για τη δημιουργία ενό ισχυρού πλαισίου που θα λειτουργεί σωστά με σαφή βήματα και ρόλου για τα διάφορα θεσμικά όργανα και του οργανισμού που θα συνεργάζονται ουσιαστικά στο πλαίσιο των διαδικασιών επανεγκατάσταση. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ απόψει όσον αφορά τι κατεξουδότηση και εκτελεστικέ πράξει, ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν στι συζητήσει μα, αλλά δεδομένη τη ε, συμφωνία για τη γενική μορφή του προγράμματο επανεγκατάσταση, δεν έχω αμφιβολία ότι θα καταλήξουμε σε λύση και εκεί υποστήριξη επίσης για τα εθνικά προγράμματα έχει συμπεριληφθεί στις τροπολογίες. Τα ζητήματα που πιστεύω θα απαιτήσουν περισσότερη συζήτηση είναι το ζήτημα των εσωτερικά εκτοπισμένων, των NDP και πώς θα συμπεριληφθούν. Οι απόψεις δίστανται μεταξύ των σκιωδών. Αυτά δεν είναι παρά μόνο μερικά παραδείγματα από τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι σκιώδεις και άλλοι συνάδελφοι ε, σε γενικέ γραμμέ θεωρώ ότι εγώ ω εισηγήτρια και μαζί με του αδελφούς μου έχουμε μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε τα πράγματα. Έχουμε διάφορε τροπολογίε που ενισχύουν ε, και μας δίνουν δυνατότητες σε εμά ω Κοινοβούλιο να παρουσιάσουμε μια έκθεση ε, στραμμένη προς το μέλλον και θετική για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και έτσι να μπορέσουμε να δώσουμε μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός οργανισμού που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα καλύτερα μέσω της συνεργασίας. Αναμένω να ακούσω τα σχόλιά σας από εσάς, τους Κιώδης και τους λίπους συναδέλφους της Επιτροπής και προσβλέπω στη συνεργασία μας ε, και στην εκπόνηση του τελικού κειμένου μαζί με εσάς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ ελπίζω να έχουμε μία αξιόπιστη πολιτική μεταγκατάσταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Δίας Δεμέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μπιόρκ για την καλή δουλειά της και για την εξαιρετική ικανότητά της να διεξάγει έναν πολύ επικοδομητικό διάλογο Έχουμε πολλές συμβιβαστικές ε, λύσεις νομίζω μπροστά μας. Οι τροπολογίες είναι αρκετά καλές ε, και αναφέρονται κυρίως σε πέντε ε, σημαντικά θέματα. Τον ρόλο των προσφύγων και της είπα της αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών από τη μία. πρέπει όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία ασύλου να συνεισφέρουν και θεωρώ πως είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ο δικός μας ρόλος, ιδιαίτερα μάλιστα από νομοθετικής απόψεως. Έπειτα, ε, ρεσιμότητα. Σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα, είμαι πεπισμένος ότι το άρθρο 4, το οποίο αναφέρει τα διάφορα κριτήρια και τις διαφορές παραμέτρους ε, που πρέπει να ακολουθήσουν ε, χώρες της Ένωσης, τρίτες χώρες και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, δεν συμφωνώ με κάτι Δεν συμφωνώ με την ε, αναφορά στο ρόλο των τρίτων χωρών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απόρριψη μιας αίτησης. Ακριβώς διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανθρωπιστική διάσταση σε περίπτωση παρατεταμένης διαμονής προσφύγων οι οποίοι έχουν περάσει αρκετά δύσκολα, έχουν διαβεβαιώσει σε δύσκολες συνθήκες. Πιστεύω ότι ο περιορισμός αυτός θα επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας αλλά και το σύνολο της κοινωνίας και θα είναι πολύ άσχημο ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Μετά, υπάρχει και η περίπτωση των ατόμων τα οποία ε, έχουν φυλακιστεί και ε, ανήκουν στις ομάδες των εκτοπισμένων. Είναι πολύ συχνά. Ε, είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εσωτερικά εκτοπισμένοι. στο Μάλι, το Ιράκ, τη Συρία, την Ιγυρία ή και την Κολομβία υπάρχει πληθυσμός εσωτερικά εκτοπισμένων αρκετά υψηλός. Στην Κολομβία, για παράδειγμα, υπάρχουν 5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι οι οποίοι είναι εξίσου ευάλωτοι και είναι εξίσου σε δύσκολη θέση με ε, τους ε, άλλους, με τους πρόσφυγες πούμε, από τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως πρέπει και αυτή η ομάδα να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Τέλος. Τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται στην πρόταση της κυρίας Μπιόρκ. Είναι κάτι που πρέπει να επανεξετάσουμε. Αναφέρονται έξι από αυτά για εσωτερικές μετακαταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως χρειάζεται προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δίας Δεμέρα. Λείπουν αρκετοί από τους κοιόδης εισηγητές, γι' αυτό λοιπόν αν θέλετε το λόγο παρακαλώ να το δηλώσετε και θα τον λάβετε. Η Σεσίλια Γουίξτρομ έχει το λόγο. Να και σήμερα επαναλαμβάνω αυτό που έκανα πριν από μερικές εβδομάδες για το ίδιο θέμα. Θα προσπαθήσω δηλαδή να εκθέσω την άποψη του σκιώδους ε, των φιλελεύθερων του Λουί Μισελ. Ο Λουί Μισελ μου έχει στείλει ένα κείμενο το οποίο θα σας το διαβάσω. Θα ήθελε καταρχάς να τονίσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και να ευχαριστήσει την Επιτροπή για την πρόταση. Το Κοινοβούλιο θα έχει τώρα την ευκαιρία να εργαστεί πάνω στην ευελτίωση των συνθήκων όσων ε, ζητούν ε, διεθνή προστασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από τους φιλελεύθερους, ο κύριος Μισελ θα περιοριστεί στο να αναφέρει τρία σημεία. Την ε, συμπερίληψη καταρχά των εσωτερικά εκτοπισμένων στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, μια που η μεταγκατάσταση είναι μια διαδικασία η οποία αφορά τους ε, πρόσφυγες που καταγράφονται σε τρίτες χώρες από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Ο κύριος Μισελ ζητά τώρα να ε, αφαιρεθούν, αφαιρεθεί αυτή η ομάδα από, το πεδίο εφαρμογής και ζητά να υπάρχει, να υπάρχει διεθνής προστασία. Μετά, Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια της δημιουργίας ενός κοινού συστήματος για το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ε, σύγχυση με την ε, νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους εσωτερικά εκτοπισμένους, οι οποίοι δεν πρέπει να υπάγονται στις ίδιες ε, διαδικασίες μετεγκατάστασης με τους υπόλοιπους. Ο κύριος Μισελ θα ήθελε επίσης να τονίσει ότι είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται βοήθεια στα κράτη-μέλη που δεν έχουν τόσο, ε, τόσο πολλές εμπειρίες σχετικά με τη μετακατάσταση και σε ό,τι αφορά τους ε, διάφορους ευρωπαϊκούς ε, φορείς και άλλους παράγοντες που ασχολούνται με την μετεγκατάσταση, ε, ο κύριος Μισελ θεωρεί πως ο ρόλος τους δεν θα πρέπει να είναι μόνο συμβουλευτικός, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να συμμετέχουν ενεργά στην ε, σύνταξη της νομοθεσίας με τις δικές του συστάσεις και προτάσεις. Επίσης, θεωρεί πως είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά η μεταγκατάσταση με τον ορισμό που της δίνει η πατιαρμοστία του ΟΕ για τους πρόσφυγες. Επίσης, σημαντική είναι και η ανταλλαγή πληροφοριών για το αποτέλεσμα της διαδικασίας μεταγκατάστασης και πρέπει επίσης να δοθεί έμφαση στην ένταξη των ε, ε, όσων μετεγκαθίστανται. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσει την κυρία Μπιόρκ για το σχέδιο έκθεσης και για την ολοκληρωμένη προσέγγισή της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Κυρία Αντζεντίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σαρτζεντίνη. Και ευχαριστώ για την ε, έκθεση, την Μάλιν. Εκτιμούμε ιδιαίτερος τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Μπιόρκ προσπαθεί να παρουσιάσει μια πρόταση που να παραμένει κοντά ε, στις αρχές των Ηνωμένων Εθνών ε, για την μεταγκατάσταση. Ε, ενώ η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη γνώμη μας, δεν αφορά τόσο τη μεταγκατάσταση, αλλά γεωπολιτικούς παράγοντες και το, τη δυνατότητα επιστροφής των ατόμων αυτών. Αναμειγνύει κίνητρα για χώρες, τρίτες χώρες που έχουν μεγάλους πληθυσμούς προσφύγων να έρθουν σε συμφωνίες μαζί μας. Και αυτό δεν πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Όσον αφορά τις προτάσεις της κυρίας Πιόρκ, οι προτάσεις αυτές είναι πολύ διαφορετικές από αυτά που προτείνει η Κομισιόν και νομίζω ότι ο τριμερής διάλογος θα είναι πολύ δύσκολος. Ε, υποστηρίζουμε το γεγονός ότι προσπαθεί να αλλάξει η ιδέα από το ένα μέγιστο αριθμό ατόμων που θα μετακατασταθούν σε έναν ελάχιστο αριθμό και ότι ε, προσπαθούμε να εισαγάγουμε σημαντικά κίνητρα για την μετακατάσταση ε, ότι παραμένουμε κοντά στα κριτήρια των Ηνωμένων Εθνών χωρίς να αναμειγνύουμε κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα ε, με το θέμα της ευαλωτότητας των προσφύγων που χρειάζονται ένα νέο τόπο για να ζήσουν να αναχαιτήσουμε την ιδέα ότι αν κάποιος έχει δικαίωμα ε, για οικογενειακή επανένωση, ότι αυτό θα πρέπει να μετράει στην ποσόστοση των μετεγκαστάσεων, βρίσκω εκπληκτικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, θεωρεί ότι αν κάποιος φέρει τον σύζυγό του ή τη σύζυγό του να ζήσει μαζί του, αυτό ε, θα μετρήσει την ποσόστοση της ε, μετεγκατάστασης. Συμπαιδεύουμε οικογενειακά θέματα με το θέμα των προσφύγων. Να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό. Ε, προτείνουμε να διευρυνθεί ο ορισμός ε, της οικογένειας όσον αφορά το δικαίωμα αυτό ε, της στα πλαίσια της μετεγκατάστασης. Αυτό που σχεδιάζουν να κάνουν οι πράσινοι είναι να υποστηρίξουν την εισηγήτρια όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάσταση που θα αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων που θα μετεγκαθίστανται μακριά από γεωπολιτικέ θεωρήσει ή άλλου είδου διαπραγματεύσει, που δεν ε, είναι προς, δεν είναι προς όφελος των ε, προσφύγων. Ε, και θα κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας για να επιτύχουμε το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Τέλος, ο κύριος Κόρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Μπιόρκ για την ε, δουλειά που πραγματοποίησε και επειδή κατάφερε να βρει τις βέλτιστες συμβαστικές λύσεις. Εμείς με τις τροπολογίες μας θελήσαμε να υποστηρίξουμε ότι ε, το εργαλείο αυτό της μετεκατάστασης είναι ένα ε, πολύ σημαντικό εργαλείο για να διασφαλίσουμε διεθνή προστασία για όλους αυτούς που έχουν δικαίωμα ε, στην προστασία αυτή. Θα πρέπει να, ε, μας, να έχουμε τα μέσα να εμποδίσουμε ε, τη δουλειά των διακινητών. Δεν θα πρέπει όμως αυτό να χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς ή σαν ένα μέσο διαχείρισης της μετανάστευσης, όπως τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ε, επ' αυτού συμφωνούμε με την εισηγήτρια όταν επιμένει στο γεγονός ότι θα πρέπει να παραμείνει ένα ανθρωπιστικό μέσο ε, η μετεγκατάσταση και όχι κάτι που συμφωνούμε με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα πρέπει να ε, ε, να μην δώσουμε στο Συμβούλιο ε, εκτελεστικές εξουσίες όσον αφορά το ετήσιο σχέδιο υλοποίησης της μετεγκατάστασης. Θα πρέπει η Κομισιόν μέσω ε, κατεξουδότηση πράξη να ασχολείται με αυτό, ε, δίνοντας αναφορά στο Κοινοβούλιο. Όσον αφορά το σχέδιο αναφοράς και τις ποσοστώσεις, μέσω των οποίων κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συμβάλλει στο πρόγραμμα κατάσταση Στην τροπολογία μας 438 ε, προτείνουμε ένα υπολογισμό που παίρνει υπόψη το συνολικό πληθυσμό, το συνολικό ΑΕΠ, ε, τον αριθμό των ατόμων που τυχάνουν ε, διεθνούς προστασίας και είναι ήδη παρόντα στο κράτος μέλος. Ε, βέβαια αυτό δεν αποκλείει τα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να διαθέσουν περισσότερες θέσεις από αυτές που προβλέπονται στο ετήσιο ε, πρόγραμμα, χωρίς αυτό να προδικάζει και τυχόν επικαιροποίηση του πλάνου πλάνου αυτού. Ε, επίσης πρέπει να δούμε τη σχέση με άλλα συστήματα όπω είναι η οικογενειακή επανένωση. Συμφωνούμε ε, επ' αυτού με την ε, εισηγήτρια ε, ότι θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιείται το μέσο αυτό μόνο όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για όλα σας τα σχόλια μα οδηγούν όλα στην ιδέα ότι χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη πολιτική επανεγκατάσταση η οποία θα πρέπει να μοιάζει με τις πολιτικές που είδαμε στον Καναδά. Όταν λέμε αξιοπιστία, να μην υπάρχει πολιτική επιρροή, να είναι μικρής κλίμακας και να χαρακτηρίζονται από ανθρωπιστική φύση, κάτι που δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια αξιόπιστη πολιτική και πιστεύω ότι πολλά από τα σχόλια που ακούσαμε και πολλέ ε, από τις τροπολογίε κινούνται προ αυτή την κατεύθυνση. Στρέφουμε τώρα στη Μάλεν για να ακούσουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα, κάποια περίληψη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ τους ε, και τους λοιπού. Υπόθηκε σαφώ από πολλούς εδώ η πρόταση της Κομισιόν απομακρύνθηκε από την ανθρωπιστική φύση και την σημερινή δομή επανεγκατάσταση όπως τη γνωρίζουμε. Και η δουλειά μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Και όταν λέω στη σωστή τους θέση και στο σωστό δρόμο, εκεί εστιάζονται οι συζητήσεις μεταξύ σκιωδών. Να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόμενοι σε υπάρχουσες δομές επανεγκατάστασης και στις σχετικές πολιτικές για να καλύψουμε τι ανθρωπιστικέ ανάγκε. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε μια ισχυρή θέση και εδώ και στου τριμερεί διαλόγου. Οι τριμερεί διαλόγοι δεν είναι ποτέ εύκολοι. Διότι εμεί στην Επιτροπή μα θέλουμε πάντα να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να ακολουθούμε κάποιε συγκεκριμένε γραμμέ περισσότερο από το Συμβούλιο ορισμένε φορέ. Όπω και να το πω αυτό, αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή έκθεση για να έχουμε μια ισχυρή θέση. Ήθελα να πω μερικά πράγματα σε σχέση με αυτά που αναφερθήκαν από τους σκεωδείς μου, ε, όπως είπαμε, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια γενική συμφωνία όσον αφορά το θέμα της αιρεσιμότητας και ότι δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή έτσι όπως την παρουσιάζει η Κομισιόν. Πρέπει να την αναδιατυπώσουμε ώστε να παραμείνει αποτελεσματικό εργαλείο ασφαλούς ε, διέλευσης ε, και για την προστασία των προσφύγων από διάφορες καταστάσεις. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για στρατηγικές απόψεις, αλλά ανά πάσα στιγμή ε, πρέπει να αναφερόμαστε στην ορολογία της υπενθυσαμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, όταν αναφερόμαστε σε τέτοια θέματα. Όπως αναφέρθηκε από πολλούς και από το Λίμισελ ε, γίνονται συζητήσεις ε, για τη συμπεριλήψη των εσωτερικά ευτοπισμένων. Ελπίζω να καταφέρουμε να βρούμε μια λύση που θα βρει σύμφωνους άπαντες Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε. Αλλά θα το συζητήσουμε στην πρώτη συνάντηση σκιωδών φυσικά. Όσον αφορά ορισμένα από τα ζητήματα που ανέφεραν άλλοι συναδελφοί περί αριθμών, όλες οι τροπολογίες για θέματα αριθμών κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ε, προς μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση και ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό. Δεν ε, σχολίασα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έγιναν πολλά σχόλια. Θα βασιστούμε στη σημερινή αρχιτεκτονική, στι σχέσει μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων και τι εμπειρίε των κρατών μελών, ώστε να καταφέρουμε να μην γίνεται διπλή δουλειά και να μην γίνονται και πολλά επίπεδα δουλειά. Να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο και να αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε. Πιστεύω ότι με τι τροπολογίε μου που έχω μπροστά μου θα τα καταφέρουμε να λύσουμε αυτή την εξίσωση. Αρκετά εύκολα μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Μάλιν που απομακρυνθήκατε από την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστούμε εσάς και τους ε, σκιώδεις. Θα ψηφίσουμε είτε 10 είτε 11 Ιουλίου. Ε, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Μπορούμε να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα μέχρι τις 11.30 για την ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες για την ψηφοφορία. Δεν θα κρατήσει πολύ ψηφοφορία, αλλά είναι σημαντική. Οπότε παρακαλώ να έχετε έτοιμε τις κάρτες σας πριν ε, από τις 11.30. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, καθίστε. Θα ψηφίσουμε. Um, Συνάδελφοι, εάν είστε έτοιμοι, θα ήθελα να σας εξηγήσω πως έχουμε δύο ψηφοφορίες. Η δεύτερη σχετικά με την Eurodac. Όσοι έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν ε, στις διαβουλεύσεις, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Δεν θα ε, γίνει λοιπόν τόσο γρήγορα η ψηφοφορία, ακριβώ για να υπάρχει ακρίβεια. Η πρώτη ψηφοφορία είναι μια, μια αίτηση από τους ε, συντονιστές. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα και στις δύο ψηφοφορίες, γι' αυτό λοιπόν θέλω την προσοχή σας. Είστε όλοι έτοιμοι, έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας. Εάν όχι, παρακαλώ να μου το πείτε τώρα, διότι είναι πολύ δύσκολες οι ψηφοφορίες και το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί ακόμα και από μία ψήφο. Αν έχετε λοιπόν όλοι τις ε, κάρτες, για να τις έχετε να το πείτε. Είναι πολύ σημαντικό να είναι όλοι παρόντες. Ένα συνάδελφος περιμένει τη δική του κάρτα, υπάρχει άλλος που περιμένει. Περιμένουμε λοιπόν το συνάδελφο, έρχεται. Έρχεται σε ένα λεπτό. Παρακαλώ μην φύγετε από την αίθουσα. Περιμένουμε τους τελευταίους συναδέλφους να έρθουν. Sorry for the delay, colleagues. I'm just going to check with all the coordinators. Συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, οι συντονιστές είναι εδώ. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Τόμας ξέρω ότι είσαι πάντα έτοιμος, αλλά θα κοιτάξουμε, θα ρωτήσουμε και τους συντονιστές. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε αν δεν είναι όλοι παρόντες. Δεν είστε έτοιμοι ακόμα. Ναι, αυτό προσπαθώ και εγώ να δω, αν είμαστε όλοι εδώ. Συντονιστές, έχετε όλα τα μέλη σας εδώ. Όχι. Ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν, για να είμαστε σίγουροι. Διακοπή λοιπόν μέχρι να φτάσουν όλοι. Εντός ολίγου. Okay, those are not the members we were waiting for. Ναι, δεν είναι όμως αυτά τα μέλη που περιμένουμε. Ας το δούμε με χιούμορ. Okay, in terms of balance, thank you, Tanya. Trying to get some balance in this committee. Right, okay. Is... Μάλιστα. Οι συντονιστέ είναι ευχαριστημένοι, είστε όλοι εδώ. Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε. Προ το ΕΛΚ κοιτάζω. Ποιο είναι συντονιστή του ΕΛΚ? Εσείς. Τόμας δεν είστε εσείς συντονιστής. Ποιος είναι? Sorry, a point of order. Ένα διαδικαστικό. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, δεν ξέρω πόσους περιμένουμε. Περιμένουμε έναν, δύο, περνάει η ώρα, έχει έρθει η ώρα να ψηφίσουμε. Πιστεύω πως δεν είναι δικό μας πρόβλημα αν δεν έχουν έρθει κάποιο, κάποιοι και πίνουν το καφεδάκι τους. Εμείς είμαστε εδώ και θέλουμε να ψηφίσουμε. Βλέπω δεν είστε τακτικό μέλος αυτής της Επιτροπής, αλλά σημειώνουμε το σχολείο σας. Συμφωνούμε όλοι, μπορούμε να αρχίσουμε. Συνάδελφοι, αρχίζουμε με την πρώτη ψηφοφορία. Μετά από αίτημα τη ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, αποφάσισα να ψηφίσουμε σήμερα την απόφαση των συντονιστών να μην στείλουν επιστολή στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αναφορικά με πιθανή προσφυγή κατά παραλήψεω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων. Η απόφαση των συντονιστών ήταν να μην σταλεί επιστολή, γι' αυτό λοιπόν ακούστε. Ακούστε συνάδελφοι, προσεκτικά. Εάν, συνάδελφοι σας παρακαλώ, εάν ψηφίσετε υπέρ ηλεκτρονικά, αυτό σημαίνει ότι στηρίζετε την απόφαση των συντονιστών να μην στείλουν επιστολή. Εάν ψηφίσετε κατά, αυτό σημαίνει ότι επιθυμείτε να σταλεί αυτή η επιστολή. Επαναλαμβάνω, αν ψηφίσετε υπέρ, συμφωνείτε με τους συντονιστές να μην σταλεί επιστολή και αν ψηφίσετε κατά, επιθυμείτε να σταλεί αυτή η επιστολή. Καταλάβαμε. Περνάμε στην ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ψήφοι παραπάνω από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, προσαρμόστε το, διορθώστε το. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψηφί υπέρ 33 κατά. Καμία αποχή. Θα σταλεί λοιπόν η επιστολή. So colleagues, move straight to the uh, Eurodac vote. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για τη Eurodac. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μακοβέη. Πρωτού αρχίσει λοιπόν η ψηφοφορία, κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τις διάφορες τροπολογίες, σύντομα. Πρώτα, η κυρία Ιντφέλντ έχει μια προφορική τροπολογία 2.35 για το άρθρο 8 παράγραφος 2α νέα επιθυμεί μια τεχνική προσαρμογή της ε, τροπολογίας της που αφορά την συμβαστική τροπολογία 7. Έχετε λάβει το κείμενο της προφορικής τροπολογίας στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε την ε, τροπολογία 235 με την τροποποίηση που ε, ζητάει η κυρία Ιντφέλντ. Δεν βλέπω αντίρρηση. Ωραία. Έπειτα, έτοιμα ονομαστικής ψηφοφορίας από την ομάδα ECR για την συμβαστική 2.6 για τις συμβαστικές 2, 6 και 11. Οι υπόλοιπε με ανάταση χειρός, εκτός αν συμφωνήσουμε να γίνει η ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Το 1 πέμπτο της ε, Επιτροπής πρέπει να ζητήσει ψηφοφορία με ανάταση της χειρός. Συμφωνείτε για το ότι οι συμβαστικές 2, 6 και 11 ε, θα γίνουν με ανάταση της χειρός. Ναι, συμφωνείτε. Τέλος. Η συγκήτρια θέλει το λόγο πριν την ψηφοφορία. Κυρία Μακοβέη, ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης και όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μακοβέη. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλα θα γίνουν ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σε μένα. Αλλάξτε παρακαλώ θέση και θα σας περιμένω. Okay, colleagues, uh, we proceed with the vote. Προχωρούμε, συνάδελφοι. Συμβιβαστική 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνατε. Συμβιβαστική 1 στη σελίδα 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1, σελίδα 5. Σας περιμένω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 στη σελίδα 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 7. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2.35. Είναι η προφορική τροπολογία που ζήτησε η κυρία Ντφέλτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Στη σελίδα 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική 2 που βρίσκεται στη σελίδα 12. Ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος ε, της ομάδας ECR. Η ομάδα ECR έχει μία ψήφο παραπάνω. Παρακαλώ διορθώστε το. Τώρα είναι εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Συμβατεί με τη συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 201. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 202. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 206. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 207. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 208. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εκρίνεται. 209. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 210. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 211. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 212 και 22 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 216. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 217. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 222. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 223. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 224. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 252. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 262. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 90. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 91. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Άρχεται ψηφοφορία. Ονομαστική είναι η ψηφοφορία. Συνάδελφοι, δεν είπα ότι είναι ονομαστική ψηφοφορία. Θα έπρεπε να το έχω πει από την αρχή, έτσι είναι οι κανόνε. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν ξανά. Ονομαστική ψηφοφορία κατόπιν αιτήματο τη ομάδα ECR για τη συμβιβαστική 11. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Πέρα. Εγκρίνεται. Να μου γίνει μάθημα λοιπόν αυτό. 2.39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.41 και 2.42 ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 2.43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.45. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη συνάδελφοι, 244 ψηφίζουμε. Τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.45. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.46. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.48. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εκρίνεται. 263. Ψηφίζουμε. 263. Πέρας. Απορρίπτεται. 265. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 266. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 267. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 268. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2,70. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2,79. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 280. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 281. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 282. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 283. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 284. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.85. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.86. Η 2.86 καταπίπτει. 2.92. Α, ψηφίζουμε. 2.92. Στη σελίδα 26 βρίσκεται η 292. Α, μισό λεπτό, περιμένετε, λέει ο πρόεδρος. Sorry, colleagues, for the pause. Συγγνώμη, συνάδελφοι, για τη διακοπή. Ήμασταν στην τροπολογία 292. Ψηφίσατε όλοι. Ε, τις ψηφοφορια ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 296. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2.97, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.98, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 300. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εκρίνεται. Τροπολογία 315. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 319. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 324. Άρχεται η ψηφοφορία. 324. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 326. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 330. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 336 και 338 είναι ακριβώς οι ίδιες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. 3.42 άρχεται ψηφοφορία. 342 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας, ψηφίσατε όλοι για αυτήν την τροπολογία. Τι, ποια είπατε, 342. Εντάξει. Θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ψηφοφορία λοιπόν για την 342. Άρχεται η ψηφοφορία. του Γερούν Λενάρς. Ε, πέρας, απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην 346 ή όχι, όχι, συγγνώμη συνάδελφοι.

Εγώ επιμένω στην 344, δεν ξέρω εσείς. Τροπολογία 344. Ε, δεν μου αρέσει καθόλου να διαφωνώ με τον Ζεράρ. Με ε, θλίβει ιδιαίτερα. Λοιπόν, 344. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μετά ερχόμαστε στην 343. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 341. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται αυτή. Και τώρα η τροπολογία 346, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 354 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 355, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 356, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 362, άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 362, πέρας. Απορρίπτεται. 363, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 364. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 373 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 375 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 378 Τροπολογία 378. Άρχεται η ψηφοφορία. 378, συνάδελφοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε τώρα πάμε στην τροπολογία 48, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απόρριψεται. 380, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, 50. Which is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και 53. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Άρχεται ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 395. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 407 και 408 ταυτόσημες άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 412 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 413 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 56 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 419 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 422. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 424. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 425. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4.26. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4.29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4.35 και 4.36 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 57 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 4-38, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 4-0, Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται 441 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 442 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 4-4-5 υπέρ. Ε, συγγνώμη, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4-4-6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 4-4-7. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. 4-4-8. Άρχεται. Πέρα. Απορρίπτεται. 4-4-9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 450. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 451. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 60 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις 62 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 69 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Ονομαστική. Επειδή ζητήθηκε από το ECR. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν υπάρχουν τρεις, Λου ε, Τροπολογία 98, συναδελφοί. Δεν έχουμε χρόνο για αστεία. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 101 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 9 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τροπολογία 107 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 108. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβεστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 915. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1, 2, 3. Άρχεται η ψηφοφορία. 123. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, ζητά ο πρόεδρος, συνάδελφοι, ξέχασα την τροπολογία 130. 130. 130 άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 130. Ψήφισαν άπαντες πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 14. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 137. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Budget. Τροπολογία 16. Αυτό είναι για άρθρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ξεκολουθούμε στα άρθρα. Είμαστε στην τροπολογία 16 της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Budget. Ah, okay. Uh, colleague, sorry. Συνάδελφοι, συγγνώμη, βλέπω τι έγινε εδώ. Νομίζετε ότι η 16 ήταν η ίδια με την 16 ε, της Επιτροπής Προπολογισμών. Συγγνώμη. Λοιπόν, για να είμαστε απόλυτα σαφεί, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Θα κάνουμε πρώτα την τροπολογία 16 και μετά την τροπολογία 16 της Επιτροπής Προπολογισμών. Οπότε ξεκινάμε με την τροπολογία 16 του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τη εισηγήτρια, συγγνώμη. Ήμουν σαφής, ε. Δεν είπα budget. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της budget. Αριθμός 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Αυτή που βρίσκεται στη σελίδα 41. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία budget αριθμών 6 στη σελίδα 42 άρχεται η ψηφοφορία. Μπορείτε να αναστενάξετε με ανακούφιση. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ονομαστική. Δύο ονομαστικές. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 35 υπέρ 10 κατά 8 αποχές και τώρα ψηφίζουμε για την απόφαση έναρξης των διαπραγματεύσεων και για την διαπραγματευτική εντολή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι, όχι, όχι, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, συνάδελφοι, δεν έχει τελειώσει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι ακόμα. Περιμένετε λίγο, συναδέλφοι. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 8 κατά, 7 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια την κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ συνάδελφοι για την υπομονή σα για αυτή τη μακρόχρονη ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες.